Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la procedura di voto sull'impatto della... Μπορούμε να αρχίσουμε με την, τον αντίκτυπο της κρίσης συμβιβασμός 1 υπέρ. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Βότι κοντράρι, Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16-17 παρόμοια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 και 25 παρόμοια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. 26, 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 27 η οποία και αρχίζει. Chiusa Πέρασε. 18 εναντί 10. Ο Μάουρο ψηφίζει υπέρ. 19 λοιπόν εναντί 10, επομένως εγκρίνεται. 28 υπέρ. Όχι, όχι, καταπίπτει, λέει ο βοηθός. 29. 29, 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40-41 απανομοιότυπες. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. 40-41 ανοίγει η ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Chiusa votazione. Πέρας. 20 κατά απορρίπτεται, 42 υπέρ. Κατά αποχές. Σας παρακαλώ 42 να σηκώνετε τα χέρια. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Όχι. Κατά πίπτη. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 52. Α, όχι. 51. 51. Ηλεκτρονική, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 62 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 64 υπέρ, κατά, Ασθενούτη απο... Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα λεπτό να ελέγξω. Bene, riprendiamo Έγινε ένα λάθο, λέει ο πρόεδρο. 73, 73 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Επί της 96 αρχίζει η ψηφοφορία. Chiusa Πέρας. Απορρίπτεται για δύο ψήφους, 22 αντί 20. 23, με το μαύρο, 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές μου φαίνεται ότι έχει απορριφθεί αλλά δεν είναι απόλυτα σαφές. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της 101. Πέρας της ηλεκτρονικής 23 κατά, 20 υπέρ, 9 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται, 107 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίνεται, 108 υπέρ, κατά, απόχες απορρίπτεται, 110 υπέρ, κατά, απόχες απορρίπτεται, 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 138. Ένα λεπτό λέει ο πρόεδρος. 138. Δεν το έβρισκα. Ευχαριστώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σύμβασμος 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. 151 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 152, 152 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. 155. Α, θέλετε. Λοιπόν, 154. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 ένδυ 23. 155 υπέρ. Κατά. 14. Συμβιβασμός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 150, 152 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. 162. 162 αρχίζει η ψηφοφορία. 162 λέει ο πρόεδρος. πέρασε Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 συμβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 176 υπέρ. Κατά. Αποχές μου φαίνεται ότι έχει απορριφθεί 177 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σύμβασμος 13 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα. 182 θέλετε ηλεκτρονικό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ελέγχουμε. Πέρας για την 182. Απορρίπτεται. 13. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 192, 1 και 2, υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτονται. 194, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 195, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 196, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200, 201, 202 παρόμοιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205-206 πανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ο κύριος Λόζιν θα ήθελε να λάβει το λόγο πριν από την τελική ψηφοφορία. Γεια, dass Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα πολύ σύντομα να επισημάνω ότι έχουμε τόσες ε, πολλές διαφωνίες ως προς την έκθεση αυτή εκ μέρους ομάδας μας που θα υποχρεωθούμε να καταθέσουμε έκθεση μειονότητας. Ωραία, ε, λαμβάνουμε γνώση της ε, δήλωσης αυτής. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δύο δεν ψήφισαν. Πέρας. Σαράντα έναντι 6 εγκρίνεται να συγχαρούμε τον κύριο Λίζεκ. Ο κύριος Λίζεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής και της ΑΦΕΤ, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για την εργασία στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Αναμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας. Διακόπτουμε για δύο λεπτά. Ο κύριος Σικόρσκι φτάνει τώρα. Dear colleague, please sit down. We are... Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καθίστε παρακαλώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαφ Σικόρσκι που είναι πρώτη φορά που προσέρχεται πρώτη φορά στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων Είστε εδώ κύριε Υπουργέ για να μας μιλήσετε για τη διεύρυνση και για τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων ε, συζητήσαμε και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Νομίζω ότι κάτι θέλετε να μας πείτε και εκ μέρους της είπα της εκπροσώπου σε σχέση με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Νοεμβρίου όπου συζητήθηκε το θέμα του Αφγανιστάν, του, της Μεσογειακής Γειτονίας και θέματα ως προς το κέρας του ελεφαντουστού, το κέρας της Αφρικής, με συγχωρείτε, θα ήθελα λοιπόν να μας κάνετε μία εισήγηση και να αρκεστείτε στα 15 λεπτά έτσι ώστε να, έχουμε, να, να προχωρήσουμε σε αποκρίσει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριε και κύριοι βουλευτές, με χαρά σας συνάντησα και το Φεβρουάριο και με χαρά ξαναέρχομαι και σήμερα να σας μιλήσω με ένα μήνα ακόμα μπροστά μας για την ολοκλήρωση της Πολωνικής Προεδρίας σε αυτή την, όπως γνωρίζετε, πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στην Πολωνία θεωρούμε ότι η λύση στα προβλήματα είναι περισσότερη Ευρώπη. Και έχουμε συμβάλει προς το σκοπό αυτό Ολοκληρώνοντα Φερρυπίν ε, τι διαπραγματεύσει για το Six Pack, την δέσμη εξφέτρων. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη Συνοδοκορυφή ε, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση για το EFSF, για την ε, διαμόρφωση της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στόχος μας είναι η Ευρώπη να γίνει πιο αξιόπιστη, πιο ανταγωνιστική και πιο ισχυρή. Και βεβαίω, η μία όψη αυτού του νομίσματος είναι η ενίσχυση τη Ευρωζώνη. Η άλλη όμω όψη πιστεύουμε είναι η διεύρυνση της κοινότητάς μας έτσι ώστε να έχουμε πιο φιλόδοξ... και να έχουμε πιο φιλόδοξες πολιτικές γειτονίας ε, και ένταξη βεβαίως αλλά και μέσω του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και ή του καταπιστεύματος για τη δημοκρατία και γενικότερα για την ε, σχέση μας με, την υπόλοιπη, με τα υπόλοιπα κράτη. Μιλήσαμε λοιπόν πριν από μερικούς μήνες ε, για την διεύρυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προοπτική της διεύρυνσης και ακούστηκε ότι αποτελεί την πηγή όλων των προβλημάτων. Η θέση μου όμως είναι τελείως διαφορετική και επιτρέψτε μου να διαφωνήσω γιατί θεωρώ ότι η προσχώρηση των 12 τελευταίων κρατών μελών συνέβαλε στην ευημερία και την ανάπτυξη και των παλαιών κρατών μελών όσο και των νέων. Ο κύκλος ε, εμπορικών συναλλαγών μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών τριπλασιάστηκε με βάση τους υπολογισμού μας και έχει συμβάλει τουλάχιστον κατά 0,5% ανάπτυξη επί του ΑΕΠ για τα παλαιά μόνο κράτη-μέλη. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να προβάλλει το αντίστροφο ε, επιχείρημα, ότι δηλαδή η αύξηση, η μεγέθυνση της αγοράς ήταν ο λόγος για τον οποίο άργησε η αναγνώριση των ε, προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι η διεύρυνση λειτουργεί ικανοποιητικά και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διατηρήσει ως μία από τις κύριες προτεραιότητες του την διεύρυνση, την περαιτέρω διεύρυνση. Έχουμε μπορέσει λοιπόν να προσδιορίσουμε το τελικό κείμενο της ε, ε, συμφωνία ολοκλήρωση των με, ε, με, την Κροατία και πιστεύουμε ότι θα το εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κροατία αποτελεί χώρα υπόδειγμα για τα Δυτικά Βαλκάνια και ασφαλώς θα συμφωνήσετε και εσείς ότι ο απαραίτητος όρος είναι, όπως διαπιστώνετε, να πληρούν τις ε, προδιαγραφές για την προσχώρηση. Ολοκληρω... Κλείσαμε δύο από τα κεφάλαια της ε, διαπραγμάτευσης ε, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, αλλά όπως γνωρίζετε θα πρέπει η Άγκυρα να πληρεί και τα κριτήρια που έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εκείνους δε που δεν μπορούν ακόμη να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τις υποσχέσεις ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης και της, ανατολικής εταιρικής, και της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης. Και έτσι με τη Σύνοδο της Βαρσοβίας αναγνωρίζουμε τις φιλοδοξίες για στενότερη συνεργασία, για ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας με τα ανατολικά κράτη και την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου. Τον Οκτώβριο, στο κύριο Κρουτσένκο είπατε πολύ ξεκάθαρα τι θέση έχετε για την κατάσταση στην Ουκρανία και ελπίζουμε η καταδίκη της κυρίας Τιμοσένκο να μην οδηγεί σε περαιτέρω ε, επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης ε, στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ότι το Κίεβο θα μπορέσει να τηρήσει την, ψυχρονή, την ψυχραιμία του και δεν θα χάσει την ιστορική ευκαιρία το καρότο λίγο πολύ τη ε, προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε κι εμείς να πείσουμε με τα επιχειρήματά μας στις αρχές της Ουκρανίας. Έχουμε μπροστά μας επίσης διαπραγματεύσεις για πληρέστατες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τη Μολδαβία και την Γεωργία. Επίση, η Ουκρανία και η Μολδοβία που έχουν προχωρήσει προ το πρόγραμμα δράση για τα θέματα τη θεώρηση διαβατηρίων, θα πρέπει, πιστεύουμε, να αποζημιωθούν για τις προσπάθειές τους. Και μεταξύ των στόχων μας, στις ε, σχέσεις με τους ανατολικούς εταίρους, έχουμε την μεταρρύθμιση της δημόσιας κατά πολέμηση διαφθορά ε, και άλλα ζητήματα τα οποία θα χειριστεί η σχετική ακαδημία που ιδρύεται στην Βαρσοβία. Ένας άλλος μεγάλος εταίρο, η Λευκορωσία. 19 Δεκεμβρίου 2010. Δυστυχώ ήταν μία κακή συγκυρία Μα είχε υποσχεθεί ο πρόεδρο Λουκασέγκο ότι θα διεξαχθεί κατά τρόπου δημοκρατικού η εκλογική αναμέτρηση. Δυστυχώ όμω δεν συνέβη αυτό και αντί να συγκεραστούν οι διαφορέ, άνοιξαν περισσότερο τα χάσματα ε, και τα προβλήματα. Ελπίζουμε όμω οι φωνέ που καλούν για περισσότερη δημοκρατία να μην σιγάσουν και εμεί και βεβαίω ε, επισύουμε τη ράβδο της ε, απομάκρυνσης και των κυρώσεων και αφετέρου προσπαθούμε με κίνητρα να προσελκύσουμε την Ουκρανία και έτσι θεσπίζουμε ένα πακέτο δημοκρατικής συνεργασίας με την Λευκορωσία που θα μπορούσε να ε, ενεργοποιηθεί όταν αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και αποδειχθεί ότι η Λευκορωσία έχει ξαναβρει το δρόμο για τη δημοκρατία. Ένα πρόγραμμα ε, πλήρες μεταρρυθμίσεων, ευρωπαϊκής στήριξης, ένα πρόγραμμα που θα αποσκοπεί στη στήριξη της ε, ε, Λευκορωσίας στον δρόμο για τη δημοκρατία και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύω ότι και εσείς θα έχετε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε στη διαμόρφωση τέτοια προσφοράς. Ταυτόχρονα θέλουμε και να στηρίξουμε την Ρωσία στην προσπάθεια για εξευρωπαϊσμό εάν το επιλέξει βεβαίως, ε, την προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι, μέσα σε μια πολωνογερμανική επιστολή, αποστήλαμε τις ε, θέσεις μας προς την ύπατη εκπρόσωπο, ενθαρρύνοντας έτσι τη Λεδιάστον, στην ανάπτυξη περισσότερο φιλόδοξων ε, προοπτικών για τη σχέση με την Ρωσία. Τα συζητήσαμε αυτά και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, η εταιρική σχέση με τη Ρωσία πρέπει να στηρίζεται σε μια επικοδομητική ε, σχέση, σε νέες ευκαιρίες και βέβαια η προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι πολύ θετική εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι η Ρωσία και η Γεωργία έχουν ακόμη πολλά ε, προβλήματα να επιλύσουν, έχουν όμως συμβάλει σημαντικά στις εξελίξεις στην περιοχή τους και με τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήρη τήρηση των συνθήκων Σέγγεν ε, για υπερσυνοριακό εμπόριο μπορούμε πιστεύω να διαπιστώσουμε όταν εξασφαλιστούν όλα αυτά ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση και έτσι μπορούμε να ε, ζητήσουμε την αναθεώρηση της, ε, του κανονισμού 1931 του 2006 για τις εμπορικές συναλλαγές, τη διακίνηση αγαθών σε ε, διασυνοριακό επίπεδο. Ε, ιδιαίτερα για την περιοχή του Καλίνιγκρατ και πιστεύουμε ότι θα μα στηρίξουν σε αυτό και οι Ευρωπαίοι και εταίροι. Θα έρθει η υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και έτσι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για το εν λόγω νομοθέτημα, ελπίζω μέχρι το τέλο τη Πολωνική Προεδρία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη συμφωνία, τη συμφωνία με την Ρωσία για τι ε, διασυνοριακέ συναλλαγέ το ταχύτερο δυνατό. Φυσικά δεν θα πρέπει, κοιτάζοντας προς το βορρά και την Ανατολή της Ευρώπης, να λησμονούμε τις εξελίξεις ε, στη Βόρεια Αφρική, που ακόμα δεν έχουν σταματήσει. Ακόμα τις τελευταίες ώρες έχουμε εξελίξει σημαντικέ στην ε, πλατεία Ταχρήρ της Αιγύπτου, του Καΐρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει το ρόλο της όπως όφιλε. Πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει και με το Ευρωπαϊκό Καταπίστευμα για τη Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, να πράξουμε περισσότερα. Θα πρόκειται δηλαδή για ένα εργαλείο το οποίο ταχύτατα θα προσφέρει τη στήριξή του, την αρρωγή του σε εκείνου οι οποίοι αγωνίζονται για τη δημοκρατική αλλαγή. Στην ε, τελευταία επιστολή που συνέταξα σε συνεργασία με τη Λέβη, άστον αναφερόμαστε στον τρόπο λειτουργία αυτού του καταπιστεύματο και μιλούμε για την θέσπιση του ως καταπιστεύματο σε διεθνέ επίπεδο σε, με συμμετοχή Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών και Θεσμικών Οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με ιδρυτική πράξη που θα υπογράψουν ε, κάποια συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ορισμένα κράτη-μέλη που θα έχουν το ρόλο του σκαπανέα στην υπόθεση αυτή και που ταυτόχρονα θα υποστηρίξουν και τα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ε, είναι η ιδέα στην οποία προσκοπούμε και βεβαίω ήθελα να παρακολουθήσω και τι συζητήσει που θα αναπτυχθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Καταπιστεύματο για τη Δημοκρατία. Επίση και εν τέλει, η Πολωνία έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην εξωτερική διάσταση τη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Βεβαίω, με ικανοποίηση καταγράφουμε τι ε, ισχυρέ τοποθετήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή. Θα πρέπει να επεκταθούν οι σχέσει μα για να περιλάβουν ε, και τη διάσταση της ενεργειακής πολιτικής στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η προοπτική της Τουρκίας μαζί με το Αζερβαϊτζάν και άλλες χώρες αποτελούν μια σημαντική προοπτική, διεύρυνση των προοπτικών για τις ενεργειακές προμήθειες και όπως υπεγράμμισα και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, πέραν του νότιου διαδρόμου θα πρέπει να ε, διερευνήσουμε και την υπόθεση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου ως υπόθεση υπογραμμίζω και όχι ως μόνη λύση ε, γιατί θα μπορούσε αυτή να ε, επαναπροσδιορίσει τις τους ενεργειακούς συσχετισμούς στην Ευρώπη και μπορεί να αποτελέσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προξενεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά προς το παρόν, συνοπτικά, ως προς τις εργασίες της ε, Πολωνικής Προεδρίας και ελπίζω ότι μπορώ να στηρίζομαι στην περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Πολυπληθείς οι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο για να έχουν χρόνο όλοι θα πρέπει να μιλήσουν, να μην υπερβούν τα δύο λεπτά. Ο κύριος Σαλαφράνκα για δύο λεπτά, συντονιστής από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ, εδώ είμαι εδώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εξ ονόματος ΕΛΚ και θα ήθελα να σας υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Στην αρχή της προεδρίας σας κάνατε ορισμένες ε, δηλώσεις και είπατε ότι η Λευκορωσία είναι για την Πολωνία, ότι η Κούβα είναι για την Ισπανία. Θα ήθελα να μας πείτε πώς σκέπτεστε επί του θέματος και κατά πόσο θα υπάρχουν κυρώσεις προς τη Λευκορωσία, εάν τα πράγματα δεν κινηθούν όπως το επιθυμούμε. Ε, επίσης, έχετε 2.600 στρατιώτες στο Αφγανιστάν και είπατε ότι θα αποσυρθούν μέχρι το 2014. Θα τηρήσετε αυτή την ημερομηνία ή θα την επεκτείνετε. Επίσης, πριν αναλάβατε το Υπουργείο Εξωτερικών ήσασταν υπουργό Άμυνας και στα πλαίσια της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας υπό τις παρούσες συνθήκες και να κάνετε έναν απολογισμό για να μας πείτε κατά πόσο ε, απομακρύνθηκαν αυτές οι προσδοκίες από την παρούσα κατάσταση. Επίσης, επειδή ε, είμαι πρόεδρος της Eurolat, θα ήθελα να μας ε, συνοδεύσετε, δηλαδή μέσα στα πλαίσια των 150 ευρωβουλευτών που θα παρευρεθούν, θα, ήθελα να ε, υπάρξει και εκπρόσωπος από από την Πολωνική Προεδρία, γιατί θα μιλήσουμε για τη συνεργασία μας με τις χώρες αυτές. Θα θέλαμε να σπείτε ε, τι γίνεται ως προς εξελίξεις ε, στη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράνκα, Ο κύριος Βιγγένιν, συντονιστής από τους σοσιαλιστές, έχει το λόγο για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά και την Πολωνική Προεδρία επίσης γιατί μια εποχή κατά την οποία όλοι μιλάμε για τις δυσκολίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κατάρρευσής της, εσείς μιλάτε για την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ολοκλήρωση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να έχουν και μέλλον οι χώρες όχι μόνο οι χώρες μέλη, αλλά και οι γείτονες να δοθεί δηλαδή ένας νέος προσανατολισμός στην δουλειά μας, ιδιαίτερα στον χώρο της οικονομίας. Έρχομαι τώρα στο πρώτο μου ερώτημα. Ανησυχούμε για κάποιες τάσεις στο Συμβούλιο που καταδεικνύουν ότι ο ενθουσιασμός για τη διεύρυνση συνεχίζει να επιβραδύνεται. Θα μπορούσατε να μας πείτε ακριβώς πού πηγαίνουμε είναι η γενική τάση για τη διεύρυνση στο Συμβούλιο. Ακόμη, πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά ε, την τοποθέτηση του Συμβουλίου για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Δεύτερη ερώτηση για την Αίγυπτο. Ε, υπάρχουν επίγουσες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα τρέχοντα γεγονότα στην Αίγυπτο, τι θα μπορούσε να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την αποκατάσταση της τάξης και τη συνέχιση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα δε σε σχέση με τις εκλογές που θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα τέλος. Αναφέρομαι στο σχόλιο σας για την εξόριξη αερίου ε, Οπωσδήποτε οι σοσιαλιστές δεν είναι ιδιαίτερα ε, θαρρυντικοί και ενθουσιώδεις για την εξόριξη από αυτά τα συγκεκριμένα κοιτάσματα. Ε, έχουμε την εντύπωση ότι είναι επικίνδυνο να εξορίξουμε από το σχιστόλιθο ε, για το περιβάλλον επικίνδυνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάφτορα. Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Είσαστε αυτός που υπέγραψε επικεφαλή στην επιστολή των πέντε σε σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα. Και πολύ καλά την πιέσατε για να προχωρήσει περισσότερο η Λέιδη Άστον στην εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας. Ποια ήταν η απάντηση που σας δόθηκε Υπάρχει, συνεχίζεται η αλληλογραφία από αυτού του θέματος. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται. Δεύτερον, Μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου είναι αξιοσέβαστο πλέον να συζητάμε την τροποποίηση των συνθήκων. Τι σχόλιο θα θέλατε να κάνετε σε σχέση με τις ρυθμίσεις της Λισαβόνας όσον αφορά την ΚΕΠΑ και ειδικότερα. Πιστεύετε ότι σε μία συνθήκη στη διαπραγμάτευση για μια συνθήκη πάλι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και κάποιους αναπληρωτές για τη, πολιτικούς για την κυρία Λέιντι Άστον. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Έτκινς. Δύο λεπτά παρακαλώ. <coughs> Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε, Υπουργέ. Δύο γενικές ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα, αναφερθήκατε στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την Αίγυπτο, αλλά έχουμε και την Παλαιστίνη και, και το Ισραήλ. Έχετε στενές σχέσεις η Πολωνία με το Ισραήλ και αναρωτιέμαι αν θα μπορέσετε να πιέσετε την Ισραηλινή κυβέρνηση να κατανοήσει τα προβλήματα που προκαλούνται από από στη Γάζα από τους επικισμούς που συνεχίζονται παρά τα ψηφίσματα του, του και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πληρωτής αλλά δεν επηρεάζει τελικά τα γεγονότα σε αυτή τη δύσκολη περιοχή του κόσμου. Σας παρακαλώ σχολιάστε το κατά πόσο η Παλαιστίνη πρέπει να γίνει αναγνωριστή σαν κράτος και τι, τι νομίζετε για την ψηφοφορία που έγινε στην UNESCO, θα προχωρήσουν τα πράγματα παρετέρω. Θέλω λοιπόν την άποψή σας για την Παλαιστίνη γενικά. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι απλή. Θα ήθελα να μου πείτε αν η Πολωνία εξακολουθεί να θέλει να μπει στο ευρώ. Ευχαριστώ κύριε Άτκινς. Ο κύριος Σούλτς τώρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, εκ μέρους των Πρασίνων στην ε, Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ και για την επισκόπηση αλλά και για την αποφασιστική στράτευση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να το υπογραμμίσω. Αναφερθήκατε σε μια πολωνογερμανική επιστολή προς την Λέδη Άστον που αφορούσε την ανατολική γειτονία και την διασύνδεση της Ρωσίας σε αυτήν. Μια νέα διάσταση, είπατε, μια νέα ανατολική διάσταση στην ευρωπαϊκή πολιτική, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι εννοείτε με τον όρο αυτό. Δεδομένου ότι η Ρωσία έχει ρητά απορρίψει τη συμμετοχή της σε μια ανατολική ε, πολιτική ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι προσπαθεί να τοποθετηθεί ως υπερδύναμη και πάλι. Πώς το κρίνεται αυτό. επίση σε σχέση με την Ουκρανία, πώς ευκαιρίες, τι είδους ευκαιρίες βλέπετε να έχει η ε, προοπτική σύναψη αυτής της συμφωνίας δεδομένου ότι έχουμε τόσα πολλά προβλήματα στην ε, Ουκρανία στην πολιτική ζωή, στην υπόθεση Τιμοσέγκο. Πώς η πιθανότητα βλέπετε να έχει η κυρία Τιμοσέγκο να αποφυλακιστεί. Το έχει ο κύριος ε, Μέιερ για δύο λεπτά από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι μας κάνετε μία εισήγηση χωρίς να λάβετε υπόψη την βαθύτατη κρίση που ε, διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Η πολιτική γειτονίας παλαιότερα αφορούσε και την κοινωνική και οικονομική συνοχή και κάθε διεύρυνση συνοδευόταν από ένα χρηματοοικονομικό πακέτο, πακέτο έτσι ώστε να ενσωματωθούν τα κράτη σωστά. δυστυχώ, κάθε διεύρυνση δεν συνοδεύεται από ένα τέτοιο πακέτο. Γι' αυτό είναι δύσκολο να φτάσουμε σε μια κοινωνικο-οικονομική συνοχή. Μιλάμε για μια Ευρώπη λοιπόν δύο ε, ταχυτήτων όπου αφήνουμε την ε, αγορά να είναι αχαλήνοτη και να δρά όπως νομίζει βαθαίνοντας την κρίση. Νομίζω λοιπόν ότι η πολιτική γειτονίας θα έπρεπε να είναι μία πολιτική εμβάθυνσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης και να μην εμβαθύνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ενός και, του ενός και του άλλου τμήματος της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί μέσα στα πλαίσια της ε, των συμφωνιών σύνδεσης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πλατεία Ταχρήρ, στην, στο Κάιρο, είχαμε 34 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ασθεναρό μήνυμα έτσι ώστε να γίνουν οι συνταγματικές αλλαγές που επιβάλλονται και να απομακρυνθεί η στρατιωτική χούντα. Ως προς τις συζητήσεις για το κοσυφοπέδιο υπάρχει η έκθεση Dirk Martin η οποία ε, μιλά για τον νυν πρόεδρο του κοσυφοπεδίου σε σχέση με ε, συγκεκριμένα εγκλήματα πολέμου. Και νομίζω ότι ως προς τη δημοκρατία της ε, Κύπρου θα πρέπει να απαιτήσουμε η Τουρκία να σταματήσει την πολιτική επικισμού στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις. Κλείνει ε, το πρώτο γύρο ο κύριος Ντανζάν, υποπρόεδρος Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο Τελαφράγκα όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Προσωπικά και ως Προεδρία είχατε διατυπώσει φιλοδοξίες ευπρόσδεκτες από το Ευρωκοινοβούλιο για την πολιτική ασφάλειας και επιχειρησιακά και από την άποψη του δυναμικού με τους εταίρους της Βαϊμάρης, στην την Ισπανία Φαίνεται όμως από 14 Νοεμβρίου ότι υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, θα έλεγα ιδεολογικό, από μια χώρα από τις 27. Δυστυχώς οι φιλοδοξίες συνεπώς δεν θα υλοποιηθούν. Άρα πώς βλέπετε ρεαλιστικά και πρακτικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι και η κρίση της Λιβύης και οι περιορισμοί δημοσιονομικοί αναγκαστικά μας οδηγούν σε αμοιβαία συνεργασία στο θέμα της άμυνας παρά τις ιδεολογικές αντιρρήσεις ορισμένων χωρών. Ευχαριστώ κύριε Ντόνζον. Το λόγο έχει ο Υπουργός. Έχει τη διάθεσή του 10 λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τη δυσχέρεια που αντιμετωπίζω, γιατί δεν είμαι ο ύπατος εκπρόσωπος, έτσι. Ε, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεσμεύομαι από την αποστολή της Προεδρίας που όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι διαφορετική. Συνεπώς θα απαντήσω σαν Προεδρία που είναι υπεύθυνη η Προεδρία βασικά για τη διεύρυνση και θα σας απαντήσω και σαν ε, Πολωνός υπουργό Εξωτερικών όταν αναφέρεστε ειδικότερα στην Πολωνία. Ο κύριος Ντόνζον έχει απαντήσει στον κύριο Ντάφου ουσιαστικά. <laughs> Όσον αφορά το θέμα της άμυνας. Η Πολωνία ήθελε να προχωρήσει πιο μακριά και γρηγορότερα, αλλά είμαστε συνονετική κοινότητα σε αυτό το θέμα και πρέπει συνεπώς να διερευνήσουμε μέχρι το έπακρο την ομαδοποίηση και τον επιμερισμό που είναι πολύ σημαντικά ζητήματα σε εποχή οικονομικής κρίσης για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Ε, ε, έχουν εντοπιστεί 15 τομείς όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα κονδύλια μας σύμφωνα με τον ε, Οργανισμό Ευρωπαϊκής Άμυνας. Λοιπόν, ξεκινάμε ανάπο... ξεκινάω ανάποδα και θα φτάσω στην αρχή. Συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο Μέγιορ ότι πρέπει να βρούμε λύσεις στην Ευρώπη των 27 και ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινοτικέ διαδικασίες και τους θεσμούς μας. Σαν Προεδρία θεωρούμε ότι είμαστε οι θεματοφύλακες των συνθήκων και των κοινοτικών μεθόδων. Άρα είμαι μαζί σας αυτό. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι είμαι και κατά της δεσπόζουσας θέσης των χρηματοοικονομικών αγορών. Ε, ρωτήσανε τον Bill Clinton τι θα ήθελε να είναι μετενσαρκωμένος και είπε ότι θα ήθελα να είμαι η αγορά ομολόγων γιατί τότε θα δέσποζα στον κόσμο, θα κυριαρχούσα. Ε, ναι, φοβάμαι λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να δανειστούμε και από αυτή την άποψη όλοι είμαστε εξαρτημένοι, διότι οι αγορές αξιολογούν την αξιοπιστία μας. Και ακριβώς γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ε, περήφανος για το γεγονός ότι στην Πολωνία, παραδείγματο χάρη, έχουμε πάρει προληπτικά μέτρα για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας. Ε, δεν υπάρχει επιδρομή, αν θέλετε, κατά του πολωνικού νομίσματος. Ε, δεν, έχει, ε, δεν έχουν υπάρξει επιπτώσεις για κανένα τραπεζικό οργανισμό στην Πολωνία. Έχουμε αναπτυχθεί κάθε χρόνο. Και παρόλα αυτά η νέα κυβέρνησή μας πρότεινε ένα δύσκολο πακέτο μέτρων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά μας. Έχουμε δαγκώσει δηλαδή πλέον τη σφαίρα εμείς, την αρπάξαμε και έχουμε εξισώσει και την ηλικία συνταξιοδότηση γυναικών ανδρών στο 67. Ε, αυτό σημαίνει ότι αυξήσαμε την συνταξιδοτική ηλικία των γυναικών 7 χρόνια. Βλέπετε πόσο μας λατρεύουν. Ε, λοιπόν, είμαστε επίσης δεσμευμένοι να ανταποκριθούμε στα κριτήρια για να μπούμε στην Ευρωζώνη. Ε, και το λέω αυτό ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε αυστηρό έλεγχο των οικονομικών μας και ναι, θέλουμε να μπούμε στο ευρώ. Είμαστε εκ της συνθήκης υποχρεωμένοι να μπούμε στο ευρώ και θα πούμε όταν είμαστε έτοιμοι και όταν η Ευρωζώνη έχει βάλει και κάποια τάξη στο σπίτι της. Διάκοψε, ο μιλητής. Κύριε Σούλτς τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, πιστεύω ότι η βάση πρέπει να είναι και σταθερή και νομικά εξασφαλισμένη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν θα επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας, ε, για την οποία έχει ομόφωνη εντολή. Το συζητήσαμε αυτό στο τελευταίο FSC και μου είπαν ότι η καθυστέρηση οφειλότανε στις επιτυχημένες προσπάθειες της Ρωσίας να μπει στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τώρα που μπήκε και έγινε μέλος η Ρωσία ε, θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι φιλόδοξο το έγγραφο το οποίο ελπίζω ότι όλοι θα επικυρώσουμε ώστε να, πλέον να ξέρουμε τι να προσδοκά ο ένας από τον άλλον. Ουκρανία τώρα. Για την Ουκρατή, Ουκρανία πιστεύουμε ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα τροποποιήσει, θα μεταλλάξει αν θέλετε την Ουκρανία, θα υιοθετήσει 60% του κεκτημένου ε, και είναι μεγάλο το τίμημα και για την Ουκρανία αλλά και για μας. Ε, προσωπικά πιστεύω στην ακαιρεότητα του διαπραγματευτικού κύκλου. Εάν διαπραγματευτούμε για αυτοκίνητα, φορτηγά, ε, όνομα προέλευσης. Εντάξει. Και από την ώρα που θα μονογράψουμε, εσείς και οι χώρες μέλη θα εξετάσουν κατά πόσο η Ουκρανία πραγματικά ανταποκρίνεται στις αρχές οι οποίες διατυπώνονται ειδικότερα στην Συμφωνία Σύνδεσης. Ε, αναφέρομαι δηλαδή στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Όμως για να, για να μπορέσει η Ουκρανία να συμμορφωθεί θα πρέπει αρχικά να συμφωνήσουμε αυτά τα πρότυπα, αυτούς τους κανόνες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας αν μονογράψουμε την συμφωνία ελπίζοντας ότι οι Ουκρανικές αρχές θα το καταστήσουν πολιτικά εφικτό όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλές διπλωματικές ενέργειες γύρω από αυτό το θέμα και θα πάω και προσωπικά στην Ουκρανία αργότερα σήμερα. Ο κύριος Άτκινς τώρα. Ο κύριος Άτκινς με ρώτησε για πιέσεις προς το Ισραήλ. Φοβάμαι ότι την ερώτηση αυτή πρέπει να την κάνετε στη Λέιδη. Άστον μπορώ να σας απαντήσω σαν Πολωνός υπουργό. Η Πολωνία αναγνώρισε την Παλαιστίνη το 1988 και ψηφίσαμε στη Γιουνέκο, όπως μας ζήτησε η Λέιδη Άστον, δηλαδή απήχαμε. Νομίζω ότι απήντησα στον κύριο Νταφ. Όσον αφορά τώρα τους πολιτικούς αναπληρωτές, ξέρω τις σχετικές συζητήσεις και τις παραμέτρους, αλλά δεν είμαι άτιμος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Προσωπικά υποστηρίζω την πρότασή σας για έναν ευρωπαϊκό κατάλογο μελλοντικά στις ευρωπαϊκές εκλογές μια λίστα, ευρωπαϊκή λίστα. Και θα τοποθετηθώ και δημόσια πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Βιγγένιν πολύ σωστά με ρωτάει για τη διεύρυνση. Λοιπόν, η Σερβία μιλάει με το Κωσυφοπέδιο και ελπίζω ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με τη Σερβία κάνουμε ό,τι μπορούμε, ενώ τις επόμενες εβδομάδες. Και ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε και το ίδιο συμβαίνει και με το Μαυροβούνιο. Η Πολωνία θέλει να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια, το ταχύτερο δυνατόν. Αίγυπτος τώρα. Η Αίγυπτος είναι η θαυμάσια απεικόνηση του γιατί χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό μηχανισμό για τη δημοκρατία, διότι όπως ξέρετε οι μηχανισμοί μας ε, προχωράνε βραδέως. Λοιπόν, οι διαδικασίες για να απελευθερώσουμε ένα κονδύλι είναι τεράστιες. Ε, χρειαζόμαστε όχι μήνες, χρόνια φορά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα αυτόνομο μηχανισμό, ένα εργαλείο, το οποίο να παρεμβαίνει γρήγορα εκ μέρους που δεν έχουν εγκριθεί από καθεστώτα σε μη δημοκρατικά κράτη. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε μια καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική αν ε, μόνο μπορούμε να καταγράψουμε επισήμως τις ΜΚΟ, διότι έτσι οι δικτάτορες μπορούν να προσδιορίσουν ποιον θα βοηθήσουμε και ποιον όχι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν αυτόνομο μηχανισμό για να μας κάνει αυτή τη δουλειά. Σας παροτρύνω λοιπόν να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε αυτό το εργαλείο, το μηχανισμό. Επίσης σημειώνω ότι οι σοσιαλιστές δεν είναι υπέρ της εξόρισης ε, σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι βεβαίω κάθε εξόριξη προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα. Κάθε νέα τεχνολογία χρειάζεται κανόνες ε, που να τη διέπουν. Αλλά σας παρακαλώ να σκεφτείτε τι θα συμβεί αν η Πολωνία αλλάξει τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικού. Αυτή τη στιγμή 96% είναι από άνθρακα και ας περάσουμε τώρα στο φυσικό αέριο ξαφνικά. Οι εκπομπές θα πέφτανε δραματικά, θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη για το περιβάλλον. Ξέρετε βεβαίως για την ισορρόπηση μεταξύ κινδύνων και ευκαιριών. Πιστεύω λοιπόν ότι η ισορροπία σε αυτή την περίπτωση είναι κατά πολύ υπέρ του ε, σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Ε, θα συμβεί αυτή η πρόοδος και η εξέλιξη, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι τεράστια η βιομηχανία ήδη στη ΣΥΠΑ και το ερώτημα είναι το κατά πόσο η Ευρώπη θα μείνει στο προσκήνιο εποφελούμενη από την τεχνολογία καθιστώντας την ασφαλή ή άλλοι πάλι θα μας ξεπεράσουν. Για το Αφγανιστάν μπορούμε να μιλήσω μόνο ως Υπουργός Πολωνός. Ήμουνα και πρώην Υπουργό Άμυνα πρωτού γίνω εξωτερικών. Λοιπόν, πήγαμε στο Αφγανιστάν σαν συμμαχία, σαν ΝΑΤΟ, θα φύγουμε το 2014. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανε... αναπτυξιακές δεσμεύσεις αναλογικά με την μείωση ε, της στρατιωτικής μας δέσμευσης. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τη δεκαετία του 90 όπου οι Αφγανοί αισθάνθηκαν εγκαταλελειμμένοι και προδομένοι. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο καλό βήμα ε, μου ζήτησε η Αστον επισκεφθώ πέρυσι το, το καλοκαίρι μάλλον Αφγανιστάν, Πακιστάν και ε, πήγα και στην ομάδα του, της Κωνσταντινούπολης για το Αφγανιστάν και πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να συμφωνήσουμε για μια εντολή, για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Αφγανιστάν το ταχύτερο δυνατόν και ε, ε, ελπίζω ότι 5 Δεκεμβρίου θα το, θα το ανακοινώσουμε στη Βόνη. Τέλειωσε ο χρόνος μου. Θα ήθελα μόνο να πω στον κύριο Σαλαφράγκα ότι η Πολωνία έχει ταπεινώσει σχέση με την Ισπανία και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι άσχετα με το ποιο είναι επικεφαλής. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Θα πρέπει να σας περιορίσω σε 1,5 λεπτό έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο όσοι το επιθυμούν. Ο, το λόγο έχει ο πρόεδρος της ε, ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Μερικές παρατηρήσεις προς την διαδικασία διεύρυνσης. Ξέρουμε όλοι ότι η Πολωνία υποστηρίζει τη διαδικασία της διεύρυνσης και το επιβεβαιώσατε και εσείς με την παρέμβασή σας και δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο και να σας υποστηρίξω διαφωνώντας ταυτόχρονα με εκείνους οι οποίοι θεωρούν πως η διεύρυνση μπορεί να είναι ο λόγος ή το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχουν αναπτυχθεί τα προβλήματα που γνωρίζουμε τώρα και άλλωστε υπάρχουν και στατιστικές, ε, στατιστικά επιχειρήματα, στατιστικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη θέση ότι δεν ευθύνεται η διεύρυνση. Πιστεύω ότι μπορούμε στο 2012 να σημειώσουμε μια κάποια πρόοδο στη διαδικασία της διεύρυνσης. Σύντομα θα έχουμε πιστεύω την Κροατία και η Πολωνία μπορεί πιστεύω να σεμνύνεται για τη συμμετοχή της στην ολοκλήρωση διαδικασίας αυτής. Έχουμε ωστόσο και άλλες χώρες στην περιοχή, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, που εν μέρη το, τα, τα, τις αναφέρατε ως υποψήφιες χώρες, ε, πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά τρόπο αμερόληπτο, δίκαιο τα επιτεύγματα και προσπάθειες των χωρών αυτών στην διαδικασία για την προσχώρηση. Η Μακεδονία, η οποία πιστεύω έχει μείνει πολύ καιρό στον προθάλαμο αναμονής για τις διαπραγματεύσεις ένταξης, η Αλβανία, το Κοσφοπέδιο, το Μαυροβούνιο πιστεύω θα πρέπει να ενθαρρυνθούν έτσι ώστε να προχωρήσουν στον ίδιο δρόμο. Και κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω εσείς προσωπικά τι είδου συμπεράσματα Συμβουλίου θα μπορούσατε να θεωρείτε ε, ικανοποιητικά για τη διαδικασία διεύρυνσης, την προοπτική διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα καταλήγοντας να σημειώσω με ικανοποίηση ότι η Πολωνία αξιοποίησε και την ευκαιρία της Προεδρίας της για να καταστήσει τη χώρα την ίδια πιο γνωστή να βελτιώσει την ε, παρουσία της στη διεθνή σκηνή. Όπου και να στεκόμασταν και να βρισκόμασταν, είχαμε μπροστά μας την Πολωνία και αυτό ήταν πολύ καλό θεωρώ. Ο κύριος Φόποντα, πρόεδρος ε, της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με τα Βαλκάνια. Κύριε Πρόεδρε, ε, απερχόμενος εισηγητή για την Κροατία, μπορώ να σα βεβαιώσω ότι θα έχουμε θετική ψηφοφορία. Είχαμε 60 ψήφους υπέρ στην ψηφοφορία για την προσχώρηση, μία ψήφο κατά, μία αποχή και άρα είναι προφανές ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό για τις ε, τελικές υπογραφές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή για τη σχέση με τη Ρωσία. Είναι δυνατόν, ε, κατά την άποψη σας, μετά τη θέσπιση του παγκόσμιου την ε, υπογραφή της συμμετοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ε, και τις γενικότερες εξελίξεις να υπάρξει νέα όθηση για συμμετοχή της Ρωσίας σε μια ενδεχόμενη συμφωνία σύνδεσης και εταιρικής σχέσης. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καλό, ε, καλή προοπτική, θα ήταν καλό να δώσουμε ένα νέο έναυσμα στη σχέση μας με τη Ρωσία. Ευχαριστώ κύριε Σφόποντα, ο κύριος Στάνοκ. Συντονιστής εκ μέρους ομάδας του Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, έχοντας ακούσει και τα όσα είπε ο κύριος Κούκαν, θα ήθελα να ρωτήσω τι γνώμη έχετε για τις ε, προοπτικέ διεύθυνση προ τα, δυτικά Βαλκάνια και δει το Μαυροβούνιο, το οποίο έχω εγώ την εισήγηση και πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τα πράγματα στους επόμενου ε, μήνε. Και πότε θεωρείτε ότι θα μπορέσει η Ελλάδα να άρει το δικαίωμα τη άρνηση κυρία που έχει ασκήσει ει βάρος της Μακεδονίας για να ξεκινήσουν πλέον οι διαπραγματεύσει, γιατί είναι τελείω γελία η κατάσταση και κανεί μα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα αυτή στο δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επίση θα έλεγα ότι είχατε μάλλον μιλούσατε μάλλον υπό την ιδιότητα του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών και όχι του Προεδρεύοντος στο Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει όμως τι είδου προοπτικές ε, επιτυχίες διαβλέπετε, επιτυχίας διαβλέπετε για τις συνομιλίες τις ειρηνευτικές στην Κύπρο που φαίνεται μάλλον να έχουν ε, σταματήσει να επιβραδύνονται και σε ποιο βαθμό μπορεί η Τουρκία να επιδείξει καλή βούληση και να ε, συμβάλλει με επικοδομητικά μέτρα όπως παραδείγματι την εκένωση και απόδοση των βαροσίων. Ευχαριστώ πολύ Μπράτνερ, συντονίστρια από τους Πράσινους, παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε και από πλευρά μας κύριε Υπουργέ. Εγώ θα μιλούσα για την Συρία μάλλον. Θα ήθελα να μιλήσω για τη Συρία που δεν αναφέρθηκε. Η κατάσταση όπως ξέρουμε είναι πολύ δύσκολη. Η Ρωσία είναι μια από τι κύριε δυνάμει που παρεμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο ασφαλεία, μεγάλη και ισχυρή χώρα. Τώρα όμω με τι διαπραγματεύσει για το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δεν, μπορείτε, δεν μπορούμε, πιστεύετε, να συνδυάσουμε τα δύο και να πούμε ότι όποιο θέλει να είναι μέλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει και να αναθεωρήσει τι θέσει του σε σχέση με τη Συρία. Δεν θα έπρεπε ε, να ασκηθεί αυτή η πίεση. Όχι τόσο ανοιχτά ενδεχομένω, αλλά εν περιπτώσει θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ο τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χειρίζεται το θέμα Συρία. Δεν θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε, αν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη λέσχη, αλλάξτε στάση. Μια άλλη ερώτηση για τη Βοσνία. στην ε, αποστολή εκεί πέρα. Βλέπω ότι έχουμε μείνει σε μια στασιμότητα και δεν υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει κάποια προοπτική για σας. Και επίσης ε, η χρηματοδότηση που διαθέτουμε, η Τινησία ξέρουμε ότι είχε πάρει 50 εκατομμύρια σαν στήριξη. Δεν θα έπρεπε αντίστοιχα να δώσουμε και στις υπόλοιπες χώρες. Εγώ είμαι υπέρβεβαιος του Ευρωπαϊκού Καταπιστεύματος για τη Δημοκρατία, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που θα διατυπωθεί ε, και που θα οργανωθεί, που θα διαρθρωθεί. Ίσως θα μπορούσαμε να ε, προσέξουμε να αποφύγουμε την μορφή του τύπου Ιδρύματος Αναλίντ που τελικά δεν έχει πάρα πολύ απήχηση στις χώρες. Ο κύριος Χατζηγιώργιο, παρακαλώ, ένα μισή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες της εξωτερικής πολιτικής στην Ένωση έχουν μεταφερθεί στην ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Άστο. Θέλω να μας πείτε ποιο ποιος είναι ο ρόλος τελικά της Προεδρίας, της εκάστοτε Προεδρίας και συγκεκριμένα τώρα της δικής σας σε σχέση με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. σε επαφές έχετε με την κυρία Άστον και πόσο σας λαμβάνει υπόψη και αν έχετε κάποια παραδείγματα να μας δώσετε για το πώς στο τέλος λειτουργεί η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ε, με βάση τα νέα δεδομένα. Η δεύτερη ερώτηση. Δεν υπάρχουν σήμερα καθόλου ανοιχτά κεφάλια στην διαδικασία ένταξης της Τουρκίας. Και ήθελα να δω αν είχατε οποιοδήποτε επαφές με όσα ενδιαφερόμενα μέρη υπάρχουν, εάν έχετε κάτι να ανακοινώσετε, που να μην δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρεί καθιονδήποτε τρόπο από τις αξιώσεις που είχε από οποιοδήποτε άλλο στο παρελθόν υποένταξη κράτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Μπροκ, συντονιστής του ΕΛΚ, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, είμαι σύντομος. Συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτηση του κύριου Υπουργού των Εξωτερικών θα πρέπει να έχουμε περισσότερη δυνατότητα να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη δημοκρατίας στις χώρες που πλήττονται από δικτατορικά καθεστώτα. Έχουμε τα χρήματα γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είχαμε λόγω τη γραφειοκρατική τάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι όνειδο για μα. Είτε πρόκειται για την ε, Λευκορωσία, είτε πρόκειται για την Νότια Αφρική, το ίδιο πρόβλημα έχουμε πάντα μπροστά μα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει νομίζω να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Και συμφωνώ, σα υποστηρίζω, στην ιδέα που προτείνεται για μια κοινοτική ε, λύση που πάλι παρεμποδίζεται λόγω της γραφειοκρατικής στάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο και πιο αποφασιστικά. Ενώ εμείς είμαστε η καθοριστική ισχύση, η καθοριστική εξουσία η οποία εγκρίνει και το προϋπολογισμό, πιστεύω ότι ε, θα ήταν καλό τα 1 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπονται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αξιοποιούνται πιο αποτελεσματικά με τρόπο πιο ουσιαστικό. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό να προχωρήσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Εκ μέρους της ομάδα μου θα σας υποστηρίξουμε και πιστεύω ότι να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριος Παλέτσικη, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για τη Λευκορωσία και συμφωνώ μαζί σας όταν μιλάμε για κυρώσεις και υποστήριξη στην κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι η τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σωστή. Τι θα γίνει όμως με την απελευθέρωση των θεωρήσεων στη Λευκορωσία. Ξέρω ότι έχουν γίνει βήματα και η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα βοηθούσε στην επικοινωνία με τη Λευκορωσία. Ευχαριστούμε κύριε Παλέτσικης. Ο κύριος Πρέντα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε δύο ερωτήσεις για δύο ζητήματα. Γιατί, όπως ξέρετε, θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για το θέμα της Ισλανδίας. Ε, υπάρχει μία διακυβερνητική διάσκεψη για τις 12 Δεκεμβρίου τι θα γίνει ως προς τα κεφάλαια τα οποία ανοίγουν, πόσα κεφάλαια θα ανοίξουν και πώς. Και ως υπουργό Εξωτερικών θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με την υπερνηστερία. Πολλά ακούστηκαν, πολλές φήμες ακούστηκαν ότι δεν μπορούν να γίνει, δεν μπορεί να επιτελεστεί πρόοδος σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματι. Είσαστε ε, αισιόδοξο ως προς αυτό το ζήτημα, δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε στη λύση του ζητήματος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λίζεκ, ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια και κανείς δεν μίλησε πολωνικά, θα το πράξω εγώ. Νομίζω ότι δεν σας εκπλήξει το ότι θα μιλήσω για τη γεωργία. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε μια έκθεση επί της ουσίας και ζητήσαμε από την ύπατη εκπρόσωπο να είναι πιο επιθετική ως προς το θέμα της ε, γεωργίας. Το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πολύ σημαντικό, όπως και η Μολδαβία και η Υπερδνηστερία. Θα πρέπει να δώσουμε τέλος αυτές τις σειράξεις. Ακόμα και οι σύμμαχοί μας οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ορισμένα ευρωπαϊκά προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Βλέπετε φως στο τούνελ, εσείς και η κυρία Άστον. Υπάρχει τρόπος να επιλύσουμε αυτές τις σειράξεις. Ε, Τέλος, το λόγο η κυρία Μπόσκουρτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις, τρεις ερωτήσεις έχουν να προς το Αφγανιστάν. Τι γίνεται ως προς την ΕΕ, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα γνωρίζετε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών των υπηρεσιών αυτών, σε σχέση με τις φυλακισμένες γυναίκες στο Αφγανιστάν και υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν θα αποφυλακιστούν. Επίσης, τι θα γίνει έτσι ώστε να ενταχθεί περισσότερο η Τουρκία σε θέματα αντιμετώπισης ενέργειας, δηλαδή στο θέμα γενικότερα της ενέργειας. Βλέπουμε ότι πολλά κεφάλαια έχουν, παραμένουν κλειστά και όχι μόνο σε σχέση με την Κύπρο, αλλά υπάρχουν άλλα κεφάλαια που παραμένουν κλειστά και δεν θα έπρεπε. θα έπρεπε να κινηθούμε προς τα εκεί ως προς τις διαπραγματεύσεις και ποια είναι η άποψή σας ως προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα σε αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να μην την αφήσουμε πίσω σε σχέση με άλλες χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Δίνουμε το λόγο στον Υπουργό μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας, δηλαδή για 15 λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν για τα θερμά του λόγια για την Πολωνική Προεδρία. Τον επόμενο μήνα θα θέλαμε η Σερβία να θεωρηθεί υποψήφια χώρα τον επόμενο μήνα και για το Μαυρομβούνιο να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ως προς τη Μακεδονία γιατί υποβλήθηκε μια άλλη ερώτηση πότε θα άρει η Ελλάδα την άρνηση κυρία της για τις διαπραγματεύσεις για το ΦΥΡΟΜ φοβάμαι ότι υπερβάλλεται ως προς τη δυνατότητά μου να επηρεάσω τα πράγματα. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Φόμποντα μίλησε για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Ε, θεωρώ επίσης ότι αυτή θα πρέπει να είναι η βάση των διαπραγματεύσεων. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να μιλάμε για μια εταιρική σχέση εξυγχρονισμού η οποία θα πρέπει να μπει σε νέες βάσεις. Και δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε και οι δύο πλευρές τι σημαίνει εξυγχρονισμός. Εμείς μιλάμε για εξυγχρονισμό της κοινωνίας ως προς την εταιρική αυτή ε, σχέση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει έτσι και να μην μιλάμε για μεταφορά τεχνολογίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Αυτό θα ήταν πολύ συσταλτική ερμηνεία. Εμείς θέλουμε να έχουμε όριμες σχέσεις με τη Ρωσία και θα πρέπει να βασιστούμε και στη δική μας έννοια περί ασφάλειας ως προς τη Ρωσία και στον τομέα της ενέργειας και στο στρατιωτικό τομέα. Και ξέρετε ότι ορισμένες γείτονες χώρες, ιδιαίτερα οι μικρότερες, εκφράζουν ανησυχίες, δικαιολογημένες ανησυχίες. Γι' αυτό στην επιστολή μας με την κάθη Άστον θεωρήσαμε ότι αυτή η προσέγγιση με τη Ρωσία εξαρτάται από τη μη προκλητική στάση της Ρωσίας σε θέματα άμυνας προς τις γείτονες χώρες. και ως προς ε, την υποθετική ε, χρήση βαλιστικών πυράβλων, όλα αυτά δεν θα ήταν καθόλου, αυτό δεν θα ήταν καθόλου επικοδομητικό, όπως υποθετικά ακούστηκε. Ως προς την Κύπρο, δεν, είμαι, δεν θα είμαι αισιόδοξο ε, ε, αν δεν επιδεινωθούν τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες, αυτό θα θεωρηθεί επιτυχία. Γιατί όπως ξέρετε κύριε Τάνοκ, εκφράστηκαν ανησυχίες για τις σχέσεις μας με την Τουρκία υπό Κυπριακή Προεδρία και η Κυπριακή Προεδρία θα πρέπει να τύχει της ίδιας μεταχείρισης όπως όλες οι προεδρίες, οι προγενέστερες. Ως προς τη Συρία και για να το συσχετίσουμε με τον ΠΟΕ, θα ήθελα να το συσχετίσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ρωσία θα ήθελε τόσο πολύ να προσχωρήσει στον ΠΟΕ, έτσι ώστε να κάνει υποχωρήσεις σε άλλους τομείς. Νομίζω ότι το εμπόριο από τη φύση του είναι ένα ε, όπλο με διπλή αιχμή και δεν νομίζω ότι ε, θα επιτύχουμε σε αυτό το τομέα. Ελπίζουμε να αλλάξει η θέση εξαιτίας του αραβικού συνδέσμου. Γιατί άλλαξε δηλαδή και ο αραβικός σύνδεσμος τη θέση του και νομίζω ότι επίσης προς τη Συρία όλο ένα και διονγκούται. Θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξο, αλλά δεν μπορώ. Ως προς το θέμα της Βοσνίας, μπορώ να σας πω ότι η Πολωνία καταβάλει κάθε προσπάθεια. Όπως ξέρετε έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις στη Βοσνία, ενώ πολύ μεγαλύτεροι πέκτες έχουν αποσύρει τη δική τους δύναμη. Επίσης και στο Κωσυφοπέδιο πεδίο υπάρχει στρατιωτική δύναμη καθώς και στην KFOR υπάρχει δική μας στρατιωτική δύναμη. Εάν και οι άλλοι έκαναν το ίδιο θα είχαμε μια πιο σταθερή κατάσταση στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη θέση της Βοσνίας και υποστηρίξαμε τη Βοσνία μέσα στα πλαίσια της υποψηφιότητας για το Συμβούλιο Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος Χατζηγεωργίου με ρώτησε σε σχέση με την σχέση μεταξύ Προεδρίας και υπάτου εκπροσώπου. Ε, ανέφερα προηγουμένως ότι νομίζω ότι δημιούργησα ένα προηγούμενο υποκαθιστώντας ε, σε μια σημαντική αποστολή και σε δύσκολο χώρο ε, την κυρία Άστον. Πακιστάν και Αφγανιστάν σας είπα ότι πήγα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να χωρίσουν τα πράγματα. Προέδρευσα επίσης σε συνεδριάσεις για το Ουσβεκιστάν και για άλλες χώρες αλλά η συνθήκη άφησε ε, την Προεδρία με επιρροή σε άλλα συμβούλαια. και με κοινή απόφαση ομοδοποιήσαμε, βάλαμε μαζί μάλλον, τις δυνάμεις μας για τις εξωτερικές υποθέσεις. Προχωρήσαμε σε κάποιες μεταβολές, μεταρρυθμίσεις και θα περιμένετε, θα μπορείτε να περιμένετε μία επιστολή από διάφορες χώρες ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες. Ως προς τη Τουρκία τώρα, ε, πολλές ερωτήσεις μου κάνατε, δεν έχω ούτε καλά νέα ούτε κακά. Χρειάζεται συνένεση, ομοφωνία και απλώς δεν υπάρχει η ομοφωνία. Αν κατάλαβα τον κύριο Μπρόκ σωστά, ναι, πρέπει να βρούμε πιο αναλυτικό τρόπο για να δαπανίσουμε τον προϋπολογισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό. Ε, η προσέγγιση δεν είναι να φτάσουμε στα κονδύλια που αναφέρατε. Η ιδέα είναι να ξεκινήσουμε από κάτι μικρό και να μεγαλώσουμε σιγά σιγά. Αν βεβαίως μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, ε, μπορεί να βρεθεί ένα παράδειγμα πώς να επιταχύνουμε τις διεργασίες, ίσως αυτό να ακολουθηθεί και από άλλου θεσμού. Ο κύριος Παλεύσκη ρωτάει για την θεώρηση, για τη Λευκορωσία. Ε, θεωριστή απατηρίων. Δηλαδή, ε, συμφωνώ με την ουσία ότι δεν πρέπει να τιμωρήσουμε το λαό της Λευκορωσίας για όσα κάνει η εξουσία. Αλλά βεβαίως το θέμα της χορήγησης θεώρησης είναι κυρίαρχο δικαίωμα μιας χώρας και συνεπώς είναι αδύνατο να παρέμβει κανείς σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, με πάση περιπτώσει, ε, χωρίς την συμφωνία της κυβέρνησης έχουμε υπογράψει και επικυρώσει συμφωνία για την κυκλοφορία μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Έχει επικυρωθεί πλήρως από την Πολωνία και νομίζω ότι το ίδιο έχει κάνει και η Λευκορωσία. Αλλά ο πρόεδρος Λουκασέγκο επικύρωσε και στην συνέχεια το βάλε στο ζυρτάρι. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα εσείς. Έκανα ό,τι μπορούσα πρέπει να σας πω. Πρώτα απ' όλα χαμήλωσα το τιμήμα, την τιμή μάλλον, και μετά κατάργησα τελείως οποιαδήποτε επιβάρυνση για την έκδοση θεώρησης για τη Λευκορωσία και έχει, η ζήτηση έχει αυξηθεί κατά 400%. Αλλά όσον αφορά τις θεωρήσεις ε, Σέγγεν, χρειαζόμαστε τη συνεργασία των ε, των ε, αρχών της Λευκορωσίας και από ό,τι καταλαβαίνω η Κομισιόν δεν έχει συναντηθεί με τη Λευκορωσία. Ε, λοιπόν, ακόμη και όταν προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί, σαν εταίρος η Λευκορωσία παραμένει δύσκολος. Διέκοψε ο μιλητής. Ισλανδία. Ναι, έχουμε ανοίξει τη διαπραγμάτευση για πέντε κεφάλαια και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε τρία σχεδόν άμεσα. Υπερδνηστερία. Πολύ καλή ερώτηση. Παγωμένη σύγκρουση που θα για την οποία θα έπρεπε κάτι να γίνει. Αν είστε κάποια δύο εδώ, Μολδαβία είναι πολύ δραστήρια σαν χώρα προχωράει με προευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις και νομίζω ότι πρέπει να να την επενέσουμε. Όσον αφορά την πρωτοβουλία Μέσενμπεργκ, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή. Θα πρέπει η Ρωσία να είναι σοβαρή στη σχέση της με την υπερνηστερία και τον κύριο Σμύρνοφ και είναι θέμα αν θέλετε, ένα τεστ ως προς τη Ρωσία, δηλαδή κατά πόσο έχει τη θέληση και την ικανότητα να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τον στρατηγικό μας διάλογο Άστον Λαμπρόφ, ε, αρκεί να υπάρχουν αποτελέσματα. Δηλαδή όχι να ανοίγουμε επισήμως ένα διάλογο, ε, κάπου πρέπει να κατατείνει αυτός ο διάλογος. Και ενώ η υπερνηστερία είναι ένα μικρό έδαφος, η αρνητική επίπτωση αποσταθεροποίησης της Μολδαβίας και της Ουκρανίας από την υπερδυνιστερία είναι σημαντική και συνεπώς χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ρωσίας και χρειάζεται να επιμείνουμε προς τις ρωσικές και ουκρανικές αρχές και στις αρχές Πρέπει επίσης να επιμείνουμε προς τις αρχές που έχουν αποσχιστεί ότι το status quo δεν είναι αποδεκτό. Κύριε Λίσεκ, συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Μακάρι να μπορούσα να είμαι αισιόδοξο για αυτές τις παγωμένες συγκρούσεις εντό εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε αυτό που θέλω να πω, ότι κάτω από τη σημερινή ηγεσία της Ρωσίας και της Γεωργίας το βρίσκω πολύ δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξο, διότι δεν είναι μόνο κράτος προς κράτος, είναι και προσωπικό. Ωστόσο, εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επαραδείγματι, η αποστολή επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται υπό την διοίκηση στρατηγού Πολωνού. Αφγανιστάν χώρα την οποία γνωρίζω καλά. Έχω ταξιδέψει επί 28 χρόνια την επισκεπτόμουν. Έχω γράψει και το πρώτο μου βιβλίο για το Αφγανιστάν. Πρέπει να σας πω ότι στο Αφγανιστάν αντιμετωπίζουμε ένα δίλημα η κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν δεν είναι σύμφωνη με τι δικέ μα προδιαγραφέ, αλλά πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε κι εσεί πω πάντω είναι καλύτερη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από ό,τι υπήρξε ποτέ στο παρελθόν του Αφγανιστάν και δει το καθεστώ ε, από το οποίο απαλλάξαμε το Αφγανιστάν, δηλαδή τον Ταλιμπάν. Υπάρχουν δύο διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις σε σχέση με το Αφγανιστάν, που θεωρώ αντιφατικές. Πρώτον, Θέλουμε να γίνονται σεβαστές οι απόψει των μειονοτήτων και των Αφγανών. Φερρυπίν, τις μείνοντα των ΣΙΑ. Από την άλλη όμως θέλουμε και τις απόλυτες προδιαγραφές που αποτελούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελεί το ζήτημα της μεταχείρισης των γυναικών. Θέλουμε αυτά όλα να ενισχυθούν. Οι Αφγανοί ίδιοι όμως και κάποιες μειονότητες του Αφγανιστάν διαφορετική άποψη. Και άρα έχουμε ένα ε, ηθικό δίλημα στο τι από τα δύο θα επιλέξουμε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οποιοδήποτε όπως εγώ έχει επισκεφθεί τη χώρα αυτή επί 25 ε, έτη μπορεί να αντιληφθεί αυτή την κατάσταση. Υπήρχαν λοιπόν πολλά προβλήματα πριν από 25 χρόνια στο Αφγανιστάν. Ήταν τελείω διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και μπορεί να υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, αλλά έχουμε σημειώσει και σημαντική πρόοδο. Σα διαβεβαιώ δε ότι όσον αφορά το θέμα της μεταχείρισης των γυναικών, η Λέδη Άστον, και την έχω δει εν δράση, είναι ιδιαίτερα ε, δραστήρια και αποφασιστική και αγωνιστική. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πολύ ε, επικοδομητική αυτή η συνάντηση. Αρχίζει ένας διάλογος ο οποίος θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Ξέρετε το ενδιαφέρον μας, το μεγάλο ενδιαφέρον μας, αλλά και την θέλησή μας να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε και θα ξαναειδωθούμε όταν θα έχουμε εξελίξεις μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Στις 11.30 υπό τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ, θα έχουμε την διάσκεψη Σαχαρόφ με τους τιμημένους των προηγούμενων ετών και θα μιλήσουμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και απόψε θα έχουμε μία θα έχουμε μία εκδήλωση στο Παλέντε Μποζάρ. Η επόμενή μας συνεδρίαση θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου στις 2 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.